Κύριε Ριβελίνη. Ευχαριστώ πρόεδρε και βεβαίω ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, συναδέλφους. Εγώ ζήτησα να υπάρχει μεγαλύτερη, να υπάρξει κάποια ανατροπή τη ημέρησης διάταξη, μόνο να αλλάξει το δικό μου θέμα με του κυρίου Μόλντερ. Δηλαδή, η έκθεση του κυρίου Κάλβιν ε, μπορεί, θα μπορούσε να έχει γίνει πριν από μένα, αλλά παρόλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, ευχαριστώ όλου ε, που είχαν την ευγενή καλοσύνη να με εξυπηρετήσουν και να προταχθεί η δική μου η έκθεση. Τώρα, όσον αφορά την έκθεση την οποία τώρα εξετάζουμε είναι ιδιαίτερα σημαντική κύριε Πρόεδρε και τούτο διότι βρισκόμαστε σε μια τέτοια χρονική στιγμή της οικονομικής κρίσης όπου η συμμετοχή των κοινοτικών ταμείων καθιστά απαραίτητη την αναθεώρηση των χρηματοδοτικών μέσων. Ο στόχος λοιπόν αυτής της έκθεσης είναι να βελτιωθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση κυρίως για όσους εκτελούν έργα έτσι ώστε οι τελευταίοι να μπορούν να έχουν πρόσβαση στα υπάρχοντα κονδύλια και για να γίνουν όλα αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να συσταθεί ένα εργαλείο επιμερισμού του κινδύνου, ένα εργαλείο το οποίο περιλαμβάνει ένα κομμάτι των κονδυλίων που δεν χρησιμοποιήθηκαν από τα κράτη-μέλη, κυρίως αυτά που προήλθαν από τα διαρθρωτικά ταμεία και σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή και ε, με άλλους ε, χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς ε, που έχουν πολιτική αποστολή, όλα αυτά τα ταμεία, όλα αυτά τα κονδύλια να επιστρέφονται. Εγώ λοιπόν προτείνω κάποιες αλλαγές και οι αλλαγές αυτές έχουν στόχο να βελτιωθεί η ε, δυνατότητα εφαρμογή αυτής της ε, πρότασης και θα μου επιτρέψεις να αναφέρω αυτές τις τροποποίησεις. Πρώτη τροποποίηση, η δυνατότητα να επεκτείνονται τέτοιου είδους μηχανισμοί επιμερισμού του κινδύνου σε όλα τα κράτη-μέλη έτσι ώστε να ισχύει η εξή αρχή καλύτερα το προλαμβάνει από το θεραπεύει. Άρα δηλαδή, αν επεκταθεί αυτή η ρύθμιση σε όλα τα κράτη-μέλη, με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να αποφύγουμε επικίνδυνα δημοσιονομικά ελλείμματα. Δεύτερη τροποποίηση δική μου. Επειδή η πρόταση θα έχει επιπτώσει στην πραγματική οικονομία των κρατών μελών, ε, όπως επίσης και στις αποφάσεις που θα ληφθούν, πρέπει ο κανονισμός αυτός να ισχύει ε, τόσο για τις ε, παρεμβάσεις των διαρθρωτικών ταμείων όσο και για την υποδομή και τη λειτουργία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που κύριε Πρόεδρε είναι ο πραγματικός πλούτος της Ευρώπης. Τρίτη πρότασή μου. Η συμμετοχή στο Ταμείο θα πρέπει να λαμβάνει χώρα με βάση τα αιτήματα μεμονωμένων κρατών μελών χωρίς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπορεί αυταίρετα και κατά τον δοκούν να εφαρμόζει την αρχή της επιλεξιμότητας. Και η τελευταία μου πρόταση είναι ότι εγώ προσωπικά πιστεύω ότι για να βελτιστοποιήσουμε αυτό το εργαλείο του επιμερισμού του κινδύνου και για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε στον ιδιωτικό τομέα την υλοποίηση έργων, για να τα πετύχουμε όλα αυτά είναι απαραίτητο οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στο άρθρο 56, ο περιορισμός αν θέλετε του άρθρου 56 να διαγραφεί, να κυρωθεί. Βεβαίως, ως Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμών, επιθυμώ η Επιτροπή αυτή να ενημερώνεται αδιάλειπτα και η Επιτροπή η δική μας να μπορεί και να ελέγχει την, ε, την χρήση των κονδυλίων και την διοχέτευσή τους, έτσι ώστε να μην προκύπτουν περιττές δαπάνες που να επιβαρύνουν τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Όπως σας λέω, αυτό που μας ενδιαφέρει ε, κυρίως και μεταξύ άλλων είναι να γίνεται καλύτερη χρήση των εκταμιευόμενων κονδυλίων. Σας ευχαριστώ κύριε Λιβελίνη. Ο κύριος Γκονσάλβες είναι παρόν από πλευρά Κομισιόν. Αν επιθυμεί να λάβει το λόγο. μόριστε. Παρακαλώ να τοποθετηθείτε εφόσον το επιθυμείτε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μας για τη γνωμοδότηση του εισηγητού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ευχαρίστως σημειώνει ότι η γνωμοδότηση του εισηγητού για την πρόταση της Κομισιόν είναι θετική. Πρόταση σημαντική σε στιγμές κρίσεως και ιδιαίτερα για τις ε, χώρες μέλη οι οποίες λαμβάνουν ενίσχυση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και δεν είναι σε θέση να ασκήσουν την πολιτική συνοχή στα διάφορα έργα. Και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι το μέτρο πρέπει να περιοριστεί στις χώρες εκείνες μέλη οι οποίες λαμβάνουν χρηματοδότηση από το Διεθνές Νομιωτικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Ένωση και αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωζώνης από τον Ιούλιο του 2011 έδωσαν ξεκάθαρα το μήνυμα στήριξης των χωρών αυτών μελών με λήψη ιδιαίτερων μέτρων που να επιτρέψουν τη χρηματοδότηση έργων συνοχής. Και το μέτρο λοιπόν αυτό συμβαδίζει με τις κατευθύνσεις που έδωσαν οι αρχικοί κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωζώνης. Εκτός αυτού η Κομισιόν δεν γνωρίζει άλλες χώρες μέλη που να έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για την εφαρμογή του μέτρου αυτού. Μόνο από την Ελλάδα έχουμε λάβει σχετική αίτηση μέχρι τώρα. Το μέτρο λοιπόν έχει σχεδιαστεί ιδιαίτερα για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση στην Ελλάδα και σε ό,τι αφορά τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογή του μέτρου σε έργα εκτός της πολιτικής συνοχή, από πλευρά Κομισιόν θεωρούμε ότι εδώ ίσως ελοχεύουν κίνδυνοι διότι η, πολιτική συνοχή η χρηματοδότηση πολιτικής συνοχής που στοχεύεται με το μέτρο αυτό απευθύνεται στην εκπλήρωση ορισμένων έργων σε ορισμένους τίτλους του προπολογισμού, του πολιετούς πλαισίου η χρηματοδότηση άλλων έργων εκτός πολιτικής συνοχής θα οδηγήσει σε νομικέ περιπλοκέ και επίση δεν θα εντάσσεται στον προπολογισμό. Σε ό,τι αφορά τι μικρέ και μεσές επιχειρήσει, ήδη έκθεση διαβιβάστηκε στον πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού για κονδύλια, για μέσα μάλλον, τα οποία είναι στη διάθεση των μικρών και μεσών επιχειρήσεων ήδη τώρα. Άνω των 8 εκατομμυρίων ευρώ και μπορούμε να κάνουμε ακόμη περισσότερα, να τα συνδυάσουμε και με δάνεια για τις χώρες οι οποίες λαμβάνουν ε, στήριξη για το εισόδημα. Δύο λεπτά ακόμα, Πρόεδρε. Στην πρόταση του εισηγητού περιλαμβάνεται μια ένδειξη ότι το μέσο αυτό μπορεί να έχει επιρροή και στη χρηματοδότηση άλλων ε, μέσων φροντίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι χώρες εκείνες που έχουν προβλήματα απορροφητικότητας να μην υποστούν ζημία. Ο στόχος μας είναι να διευκολυνθεί η χρηματοδότηση της πολιτικής συνοχής στις χώρες μέλη όπου δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν τώρα τέτοια έργα, διότι ο ιδιωτικός τομέας δεν μπορεί να συνεισφέρει τα απαραίτητα κεφάλαια. Δεν είναι λοιπόν μέτρο διευκόλυνση της απροφητικότητας. Τέλος, αναφέρω ότι για να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εφαρμόσει το μέτρο αυτό υπό κεντρική διαχείριση, παίρνει χρήματα από την κοινή διαχείριση για να γίνει η απευθείας διαχείριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή άλλη δημόσια τράπεζα. Αυτό όμως για να γίνει αυτό θα είναι απαραίτητο τα μέσα αυτά να είναι εξαιρετικά περιορισμένα σε ό,τι αφορά το πεδίο εφαρμογή του και δεν θα είναι δυνατόν κατά κάποιο τρόπο να σχεδιαστούν τα μέτρα στα μέτρα των διάφορων χωρών μελών. Πρέπει να λοιπόν να παραμείνουμε στα πλαίσια των διευρωπαϊκών δικτύων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κύριε Κονσάλβες. Τρεις συνάδελφοι τώρα ζητούν να λάβουν το λόγο. Ο κύριος Χάρτουγκ. Από όσο κατάλαβα, ο στόχος είναι περισσότερα κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να εισρεύσουν σε χώρες μέλη, από αυτές που βρίσκονται στο τέλος της σειράς. Οι τράπεζες δεν θέλουν να δώσουν λεφτά, οι χώρες μέλη δεν, δεν θέλουν πια να δώσουν λεφτά, τα διαθωτικά ταμεία και τα Ταμείο Συνοχής επίσης δεν θέλουν πια να δώσουν χρήματα και διαρωτώ με, μήπως έχουμε τρελαθεί και πάμε να του ρίξουμε και άλλα μέσα, και άλλα λεφτά. Ο Πρόεδρος, σα ευχαριστώ. Ο κύριος Σταυρακάκη. Thank you very much, Mr. Chairman. Dear colleagues, from my side... Από τη δική μου πλευρά, χαίρομαι για το σχέδιο γνωμοδότησης. Ο κύριος Ριβελίνη νομίζω ακολουθεί τη σωστή πορεία. Στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης το συζητήσαμε το θέμα διεξοδικά και θεωρούμε ότι η Κομισιόν έχει υποβάλει σωστή πρόταση και αυτή έχει μεγάλη σημασία να επιτευχθεί δηλαδή συμβασμός όσο το δυνατόν ταχύτερα. Για να επιτύχει η πρόταση το στόχο της είναι σημαντικό να κινηθούμε γρήγορα. Μόνο τότε θα έχουμε το δυνατόν περισσότερα θετικά αποτελέσματα επί από Αυτά δηλαδή που στοχεύει η πρόταση. Όσο περισσότερες καθυστερήσει σημειωθούν, τόσο λιγότερο θα είναι το αποτέλεσμα. Δύο σχόλια και δύο τροπολογίες. Πρώτο, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι είναι σαφές ότι το μέτρο επιμερισμού, το μέσο επιμερισμού συμβαδίζει με τη στρατηγική του 2020, διότι εξυπηρετεί ευρύτερου στόχους από αυτούς του ERDF, τη ε, Περιφερειακής Ανάπτυξης δηλαδή. Τε, δεύτερο σημαντικό είναι ο ρόλος των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, που είναι ραχοκοκαλιά της οικονομίας της Ένωση, και που αυτές μπορούν να οδηγήσουν ξανά στην ανάπτυξη με την δημιουργία απασχόληση και καινοτομία. Ναι, μεν χρειάζεται αύξηση τη χρηματοδότηση των μικρών και μεσών επιχειρήσεων. Η γνώμη μου είναι ότι τα υφιστάμενα χρηματοδοτικά μέσα ενισχύουν την λειτουργία των μικρών και μεσών επιχειρήσεων και επομένως θα αυξήσουν και τη ρευστότητα. Ωστόσο, υπάρχει κίνδυνος εδώ να πέσουμε σε επικάλυψη ή να ακυρώσουμε άλλα μέτρα εφαρμογής. Ευχαριστώ. Ιβάνοβα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή μας για την πολύ καλή δουλειά που έκανε και επίσης ε, θα ήθελα να χαιρετήσω και την πρόταση επιτροπής ε, που προβλέπει την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, την ενίσχυση ε, των κονδυλίων των διαρθρωτικών ταμείων. Νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσουμε ότι η χρηματοπιστωτική κρίση είναι ε, συστημική. Δεν πλήττει μόνο ένα κράτος μέλος. Και ε, πρέπει να έχουμε μια ολιστική προσέγγιση ότι υποφέρουν όλα τα κράτη-μέλη και όταν υπάρχει ε, δημοσιονομική στενότηση ε, χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ρευστότητα. Όλα τα κράτη-μέλη ε, χρειάζονται μεγαλύτερη ρευστότητα. Θα ήθελα λοιπόν να διευκρινίσω το εξή. Ορισμένα κράτη-μέλη καταβάλουν τεράστιε προσπάθειε για να διατηρήσουν τη δημοσιονομική πειθαρχία και να περικόψουν τι δημόσιε δαπάνε. Γιατί να μην επιτρέπεται σε αυτά τα κράτη να έχουν την ίδια πρόσβαση στο εργαλείο αυτό. Ε, αλλιώς δίνουμε λάθος μήνυμα, εκπέμπουμε λάθος μήνυμα που θα οδηγήσει ε, στο ότι ορισμένα κατημέλη θα αγνοήσουν ε, το τι κάνουν οι υπόλοιποι και θα προχωρήσουν στο δικό τους δρόμο, πράγμα που θα ήταν αρνητικό. Θα θέσω κάποιες δικές μου τροπολογίες, θα υποβάλω κάποιες πρωτολογίες και ελπίζω η Κομισιό να αναθεωρήσει τη θέση της. Πρόεδρος, ε, δεν βλέπω να έχει ζητήσει κάποιος άλλος το λόγο, δεν ξέρω πως ο εισηγητής επιθυμεί να επανέλθει. Ναι, Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για όλα αυτά που είπαν και θα μου επιτρέψετε κάποιες διευκρινήσεις. Καταρχήν απευθύνομαι προς τον κύριο Χάρτουμ. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι δεν προβλέπετε καμία αύξηση δαπανών. Ε, κάθε άλλο, απλά με την πρότασή μου ε, προβλέπω καλύτερη χρήση των ήδη υπαρχόντων κονδυλίων, όχι να αυξηθούν οι δαπάνες. Δεν καταλαβαίνω. Πού βρήκατε εσείς αυτή την αύξηση των δαπανών. Και μόνο αυτό λέω με τα ίδια χρήματα να υπάρξουν περισσότερες επενδύσει. Επουδενή λοιπόν αύξηση των δαπανών και συμφωνώ απόλυτα και με το θέμα του χρονισμού. Ε, να γίνουν όλα την κατάλληλη χρονική στιγμή. Γιατί αν υπάρχει κάτι σωστό που γίνεται άκερα, τελικά αυτό το σωστό μετατρέπεται σε λάθος. Άρα δηλαδή πρέπει να επιταχύνουμε κατά πολύ αυτή τη διαδικασία και από αυτού συμφωνούν όλοι. Ε, ευχαριστώ τη συνάδελφο κυρία Ιβάνοβα. Πράγματι πρέπει σε όλα τα κρατημέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δώσουμε την ίδια δυνατότητα γιατί η κρίση δεν πλήττει μόνο ένα μέρος Ευρώπη. Ευρώπης. Να υπάρχει λοιπόν αυτή η δυνατότητα, επαναλαμβάνω, χωρίς καμία αύξηση δαπανών με μοναδικό στόχο βελτίωση και ουσιαστική χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Αυτό πρέπει να προσφέρεται σε όλα τα κράτη-μέλη. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Ριβελίνη. Η διορία για την κατάθεση τροπολογιών είναι 14 Φεβρουαρίου του 12. Έτσι λοιπόν ε, μπορούμε τώρα να κλείσουμε το σημείο υπαριθμών 7 που είχαμε προτάξει και επανερχόμεθα στην κανονική μας ημερήσια διάταξη. Είναι ε, το σημείο υπαρτιμών 5 έκθεση Κάλφιν και εδώ καλούμεθα σήμερα να ψηφίσουμε για το σχέδιο γνωμοδότησης και θα ήθελα να δώσω το λόγο ε, καταρχήν στον εισηγητή, στον κύριο Κάλφιν. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, δεν έχω και πάρα πολλά να σας πω. Συζητήσαμε για την έκθεση αυτή παλαιότερα στην Επιτροπή μας Αναφέρουμε προφανώς την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου. Είχαμε μια πολύ καλή συζήτηση σχετικά με την αρχική έκθεση και στην Επιτροπή μας, ε, στην ε, Επιτροπή ε, Ανάπτυξης που είναι η επί της ουσίας αρμόδια Επιτροπή καλούμεθα να, να καταθέσουμε σχέδιο γνωμοδότησης ε, και θέλω τις ε, απόψεις σας. Βλέπετε ότι σε κάποια σημεία δεν είναι σαφής ε, η ορολογία και γι' αυτό λοιπόν προτείνω το εξής. Καλή είναι η έκθεση σε γενικές γραμμές και γι' αυτό για άλλη μια φορά ευχαριστώ στους αδέλφους που κατέθεσαν πολύ χρήσιμες παρατηρήσεις. Πρόεδρος, αν λοιπόν συμφωνείτε να ξεκινήσουμε με την ψηφοφορία που είναι εν μέρη ηλεκτρονική. Το λέω αυτό για να προετοιμαστείτε ως προς τις ε, κάρτες σας. Ε, πάμε λοιπόν στην ε, τροπολογία υπαριθμών 1. ψηφίζουμε σε τμήματα. Τροπολογία Bath Styles. Παρακαλώ, ποιος είναι υπέρ του πρώτου τμήματος. Ναι, το χέρι κατά. Αποχές ε, οριακό το αποτέλεσμα. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Υπέρ παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Έκλεισε. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Ψηφίζουμε για το δεύτερο τμήμα. Υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Κατόπιν παράγραφος 3α, ε, τροπολογία 2, υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται και αυτή τα τροπολογία υπαριθμών 3 υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 4 υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 5 Ρολάντας Πάξας υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 6. Εδώ παρακαλώ, παρακαλούμε ηλεκτρονικό έλεγχο για την προηγούμενη την υπαριθμών 5. Ψηφίζουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Τροπολογία υπαριθμών 5. Ε, έκλεισε παρακαλώ η ψηφορία. Το αποτέλεσμα. Απορρίπτεται. Τώρα, τροπολογία υπαριθμών 6. stops. Υπάρχει προφορική ε, τροπολογία. Ψηφίζουμε λοιπόν υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία υπαριθμών 7. Ψηφίζουμε σε τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, υπέρ, κατά, για το υπόλοιπο ψηφίζουμε τώρα αποχές, απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για το δεύτερο τμήμα. Ε, υπέρ παρακαλώ. Ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Πάμε στην τροπολογία 8 με προφορική τροπολογία. Υπάρχει κανείς που να διαφωνεί με αυτή την προφορική τροπολογία. Όχι ψηφίζουμε. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Κατόπιν. Τροπολογία υπαριθμών 9. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Έτσι ε, ψηφίζουμε τώρα ε, για το σύνολο του σχεδίου γραμματότησης ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Ε, 20 υπέρ, 2 κατά, καμία εποχή εγκρίνεται. Πάρα πολύ ωραία και ευχαριστούμε και τον εισηγητή και έτσι κλείνει και αυτό το θέμα της ε, ημερήσιας διάταξης και πάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, το 6. που είναι η αντιπροσωπεία στην ΑΙΤ. Ε, να δώσω το λόγο στον κύριο Μούλντερ. Κύριε Μούλντερ, έχετε το λόγο. Ε, πρόεδρε, θα είμαι πολύ σύντομος. Ε, είχαμε ε, πάρα πολλές ε, συζητήσεις για να προετοιμάσουμε αυτή τη συνάντηση στην ΑΕΤ. Είχαμε μία ενημέρωση για την κατάσταση ασφάλειας και νομίζω είχαμε και μία συνάντηση με έξι ΜΚΟ που δραστηριοποιούν στην ΑΕΤ σχετικά Σχετικά με την κατάσταση στην ΑΕΤ, η κατάσταση είναι δύσκολη εκεί. Η κυβέρνηση δεν είναι ιδιαίτερα ισχυρή. Ε, πολλοί εξ αυτών δεν είναι ιδιαίτερα στρατευμένοι στην υπόθεσή τους και όλα αυτά δημιουργούν κάποιο πρόβλημα. Στα χαρτιά σας λοιπόν, στο φάκελο, που σας έχει διανομηθεί θα βρείτε πάρα πολλές πληροφορίες για την IT. Ε, δεν μπόρεσα να διαβάσω όλες αυτές τις πληροφορίες, μπορέσατε εσείς, δεν ξέρω. Υπάρχει ένα πράγμα όπου δεν το κατάλαβε καλά η αντιπροσωπεία. Πρόκειται για την επίσκεψη της αντιπροσωπείας σε, σε τρία σημεία. Όταν συναντηθήκαμε με τις ΜΚΟ το συζητήσαμε αυτό αλλά δεν είχαμε αρκετές πληροφορίες και γι' αυτό θα θέλαμε να γνωρίζουμε ε, πώς ακριβώς γίνεται η χρηματοδότηση αυτών των προγραμμάτων. Στη σελίδα υπαριθμών 3 του προγράμματος ε, για την IT ε, υπάρχει μία πρόταση να πάμε στο ταμπάρ ίσα που περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χορηγήσει 5 εκατομμύρια ευρώ. IFRC κέντρο για την αξιολόγηση κινδύνων. Αυτό να επισκεφτούμε 5 εκατομμύρια και Σάντα Μάρς όπου πάρα πολλοί άνθρωποι ζουν μπροστά στο κατεστραμμένο προεδρικό παλάτι. Η συμβολή της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης 2,3 εκατομμύρια ευρώ. Άρα λοιπόν πρέπει να ληφθεί μια απόφαση, ε, πρέπει να αποφασίσουν οι ενδιαφερόμενοι πού θα πάνε τελικά. Αυτά κύριε Πρόεδρε για την IT θα είναι μια επίσκεψη δύο ημερών. Το πρόγραμμα είναι πολύ γεμάτο και θα δούμε τι επιτόπου, τι θα ανακαλύψουμε. Ε, δύο μέρες δεν φτάνουν για να έχει κανείς έτσι μια σφαιρική εικόνα, αλλά εν πάση περιπτώσει ε, θα αποκομίσουμε έτσι μια πρώτη ιδέα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, λέει ο Πρόεδρος, ευχαριστούμε κύριε Μούλντε και τώρα ε, θα προβούμε σε ανταλλαγή απόψεων. Και θα ήθελα να σας επισημάνω ότι το, την έκθεσή σας τη συνοδεύει μια εμπεριστατωμένη έκθεση και ε, οι αρμόδιοι εδώ στο Κοινοβούλιο ε, είναι στη διάθεσή σας για να τους υποβάλλετε ερωτήσεις. Ο κύριος Οντί ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ και την γραμματεία για την οργάνωση. Έχω τρία σχόλια. Πρώτο για την επιλογή των έργων που πρόκειται να ελεγχθούν. Συνήθως ο ελεγκτής επιλέγει κατά τρόπο τυχαίο. Εδώ τα δείγματα μας δίνονται, μας παραχωρούνται από τις υπηρεσίες της Επιτροπές. Ποιος μας λέει ότι δεν μας υποβάλλουν έργα όπου δεν υπάρχει καταρχήν κανένα πρόβλημα. Εγώ λοιπόν διερωτώ με σχετικά με τη μεθοδολογία αυτή που επιτρέπει μια πρώτη επιλογή. Λέει ότι υπάρχει θέμα ασφαλείας για τη μετακίνηση επιτόπου, αλλά παρόλα αυτά θέλω να κάνω αυτή την παρατήρηση. Δεύτερο, σύμφωνα με τις πληροφορίε που έχουμε λάβει από μη κρατικού οργανισμούς, είναι σαφές ότι για τη δημόσια αυτή χρηματοδότηση έχουν σημειωθεί σημαντικές ε, περιπτώσεις απάτης και διαφθοράς. Δεν ξέρω πώ θα μπορέσουμε να αξιολογήσουμε το θέμα αυτό τη διαφθοράς και τη απάτη, Βρισκόμαστε εν προκειμένου στην περίπτωση μιας χώρας που λόγω και της ε, καταστροφής, λόγω και της ε, δι... κατάστασης διοίκησης, δεν υπάρχει διοίκηση δηλαδή. Τρίτο σχόλιο, η Επιτροπή Αναπτύξεως του Κοινοβουλίου μας μεταβαίνει συχνά στην ΑΕΤ για λόγους που δεν έχουν απαραίτητα σχέση με τον έλεγχο προπολογισμού. Ήθελα να μάθω αν οι δύο γραμματείες έχουν συντονιστεί ώστε να έχουμε και τα έγγραφα της Επιτροπής Αναπτύξεως και αν η Επιτροπή Αναπτύξεως μπορεί να μας υποβάλει την αξιολόγηση που κάνει σχετικά με το τι μπορούμε εμεί να πράξουμε από άποψη ελέγχου του προπολογισμού. Δηλαδή, με δύο λόγια, να υπάρχει ένα συντονισμό των προσπαθειών των δύο επιτροπών. Ο πρόεδρο, ευχαριστώ. Ίσως μπορεί να απαντηθεί το ερώτημα μετά. Η κυρία Ερτσόκ. Α, κάποιο είχε ζητήσει το λόγο. Δεν πρόσεξα ακριβώ. Νομίζω, κυρία Ερτσόκ. Ο κύριος Χάρτονγκ. Δεν μπορούσα να διαβάσω σωστά το, το όνομά σας, με συγχωρείτε. Ο κύριο Χάρτονγκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ πάντοτε τα υπέρ των ελέγχων. Βρίσκω ότι είναι σωστή η διαδικασία για να γνωρίζουμε πού διοχετεύονται τα χρήματα των φορολογουμένων. Όμως, ειδικά το ταξίδι αυτό το θεωρώ ότι δεν είναι ιδιαίτερα χρήσιμο. Χθες κοίταξα μέσω του διαδικτύου τον τρόπο με τον οποίο ε, δαπανώνται τα χρήματα στην IT. Έλαβα πάρα πολλές πληροφορίες από το διαδίκτυο περί IT, άρα μπορεί κανείς να αντλήσει πάρα πολλά ε, στοιχεία από το διαδίκτυο και νομίζω ότι το ταξίδι αυτό με διήμερη παραμονή δεν πρόκειται να δώσει περισσότερα στοιχεία από όσα ήδη μπορούμε να βρούμε στο διαδίκτυο. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και το κόστος του ταξίδιου αυτού και να διαρωτηθούμε εάν όντως η ωφέλεια είναι πραγματική. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ. Δεν έχω άλλους συγκεκριμένου. Το ερώτημα λοιπόν που τίθεται τώρα είναι κατά πόσον λαμβάνουμε πληροφορίες από την Επιτροπή Αναπτύξεως Μπορεί να απαντήσει η γραμματεία. Ορίστε. Απαντώ στον κύριο Οντή. Όντως, διαβουλευτήκαμε με την ε, Επιτροπή Αναπτύξεως όχι τόσο πολύ για το πρόγραμμά μας, διότι οι αρμοδιότητες τους είναι διαφορετικές, αλλά κυρίως για πτυχές οργανωτικές και ασφαλείας. Ναι, αλλά πάντως έχουμε συνεργασία ε, στενή μαζί τους. Ο Πρόεδρος, σας ευχαριστώ. Ίσως απαντήθηκε η ερώτηση. Έχετε και άλλη ερώτηση κύριε σχετικά. Ναι και όχι. Από αυτά που ακούω από άλλους βουλευτές, οι βουλευτές της Επιτροπής Αναπτύξεως δεν γνώριζαν τα περί της δικής μας μετάβασης και εμείς δεν γνωρίζουμε τι κάνουν δεν έχω αντίληση ότι ως αξιωματούχος έχετε ε, καλές ε, επαφές μαζί τους, αλλά θέτω αυτό το θέμα ως παρένθεση αν θέλετε. Ο Πρόεδρος. Από τη δική μας γραμματεία ενημερώθηκε η γραμματεία της Επιτροπής Αναπτύξεως. Τώρα κατά πόσον ο αρμόδιος εκεί ενημέρωσε ε, την Επιτροπή Αναπτύξεως αυτό διαφεύγει των γνώσεών μου υποθέτω ότι πάντως έχουμε ανταποκριθεί στις υποχρώσεις μας. Σε ό,τι αφορά τώρα τη μετάβαση αντιπροσωπιών, ασφαλώς το θέμα της ε, αιτιολόγησης. Αυτά πρέπει βέβαια να θεμελιωθούν και ενώπιον των αρμοδίων οργάνων. Το θέμα ίσως είναι καλύτερα να τεθεί ενώπιον άλλων οργάνων ενδεχομένως και στις πολιτικές ομάδες. Από τις εμπειρίες που έχω από την Επιτροπή Περιφερειακής Αναπτύξεως μπορώ να πω ότι τα ταξίδια των αντιπροσωπιών αυτών και εφόσον είναι υπερπόντια ιδιαίτερα σημαίνει ότι πρέπει να εμβολιαστούν πρώτα οι συνάδελφοι ε, σημαίνει και μια ε, επιβάρυνση, σωματική επιβάρυνση πάντως πάντα προσφέρουν τη δυνατότητα διαφορετικής ενημέρωσης και με απευθείας συζητήσεις με τους ε, ενδιαφερομένους, δηλαδή με τρόπο διαφορετικό από την ενημέρωση που μπορεί να γίνει είτε στη βάση εγγράφων είτε μέσω του διαδικτύου. Γι' αυτό τον λόγο άλλωστε κάνουμε αυτές τις ε, προσπάθειες και θα ευχαριστήσω και είμαι, μάλλον ευγνώμων σε όλους τους συναδέλφους οι οποίοι δέχονται να αναλάβουν την προσπάθεια αυτή και τον κόπο αυτό για να μεταβούν στην ΑΕΤ. Ο κύριος Στάς. Κοιτάξτε, θα ήθελα να αφαιθώ λιγάκι σε αυτά που είπε ο συνάδελφος κύριος Χάρτουγκ. Οι επισκέψεις των αντιπροσωπιών, κατά την άποψή μου, είναι και χρήσιμες ε, και σωστές. Εγώ προσωπικά ε, επισκέφτηκα την πρώην <laughs> Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και ήταν πάρα πολύ χρήσιμη η επίσκεψη αυτή. Το θέμα είναι όμως τι γίνεται μετά με αυτές τις πληροφορίες που συλλέγαμε. Μιλήσαμε με τους ανθρώπους επιτόπου, μιλήσαμε με τα Ηνωμένα Έθνη και μετά την έκθεση της αντιπροσωπείας ε, συντάξαμε μία έκθεση ε, για να υπάρχει ένα σημείο αναφοράς. Κατόπιν τούτου συμφωνώ με τον συνάδελφο κύριο Χάρτουγκ ε, και θεωρώ οι μετέχοντες σε αυτή την αντιπροσωπεία θα συμφωνήσουν μαζί μου ότι αυτές οι δύο μέρες δεν φτάνουν. Ε, το ταξίδι είναι μακρύ και στις δύο μέρες ε, δεν προλαβαίνει κανείς να μάθει πολλά πράγματα. Ως Επιτροπή Ελέγχου του Προεπολογισμού ε, πρέπει να επισημάνουμε στο Κοινοβούλιο ότι αυτές οι σύντομες εκθέσει θα πρέπει να είναι περισσότερο με σχολή, θα πρέπει να είναι περισσότερο η εξαίρεση. Εντάξει λέει ο Πρόεδρος και θα ήθελα να δώσω το λόγο, αν το επιθυμεί βέβαια, η Επιτροπή. Θα ήθελα να καλωσορίσω την κυρία ή τον κύριο Περνασλάντο, δεν ξέρω λέει ο πρόεδρος. Με συγχωρείτε, έκανα λάθος. Η κυρία Αντριάσεν θα λάβει το λόγο λέει ο πρόεδρος. Παρακαλώ κυρία Αντριάσεν. Euh, Σας ευχαριστώ να επανέλθω στο θέμα της δειγματοληψίας των έργων. Η αφετηρία για την αντιπροσωπεία ήταν να λάβει ένα συνολικό κατάλογο των έργων που ε, αυτή τη στιγμή εκτελούνται στην ΑΕΤ και αυτό μετά από αίτημα των βουλευτών. Νομίζω ότι είναι δύσκολο για την αντιπροσωπεία να στοχεύσει σε έργα τα οποία ε, ίσως προσθέτουν κάποια αξία στην επίσκεψη χωρίς να υπάρχει κάποια παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αφενός είναι θέματα ασφαλείας, αφετέρου είναι και θέματα ε, διαρκείας των μεταβάσεων, γιατί υπάρχουν πολλά έργα τα οποία είναι στα περίχωρα του Πόρο Πράνς και η μετακίνηση από το κέντρο του Πόρο Πράνς μέχρι τα περίχωρά του, η μετάβαση αυτή λοιπόν δεν είναι ε, αυτονόητη, είναι αρκετά μακρά Γι' αυτό προσπάθησε η Επιτροπή να επιλέξει έργα τα οποία να είναι γεωγραφικά συγκεντρωμένα, διότι αλλιώς δεν θα ήταν δυνατόν να γίνουν αυτά τα πράγματα επιτόπου, δηλαδή να προλάβει η αντιπροσωπεία να τα δει όλα αυτά. Θέλαμε η, η, αντιπροσωπεία να έχει τη δυνατότητα να εξετάσει τα έργα αυτά από κοντά, γι' αυτό το λόγο ζητήθηκε από τις ε, αρμόδιες ε, υπηρεσίες να συμβάλλουν σε μια προσπάθεια προσανατολισμού περισσότερο γεωγραφικού. Όχι να αποφύγουμε να δείξουμε έργα τα οποία είναι ε, ενδεχομένως ε, ε, ε, άνευ προβλημάτων. Και γενικότερα για την Επιτροπή Συνεργασίας και Αναπτύξεως έχουμε παράσχει ορισμένα στοιχεία ενημέρωσης τα οποία περιλήφθηκαν στο γενικότερο φάκελο για να δώσουν περισσότερα στοιχεία σχετικά με την ανταπόκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ανάγκες του ε, πληθυσμού της ΑΕΤΗΣ μετά από τον ε, σεισμό. Και θα βρείτε περισσότερα στοιχεία στο ίδιο το φάκελο. Σας ευχαριστώ για τις εξηγήσεις σας, λέει ο Πρόεδρος, και το επαναλαμβάνει στα γερμανικά. Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι κλείνει εδώ ο, ο κύριος Μίλτερ. Äh, äh, Κύριε Μούλντερ, κοιτάξτε, μπορούμε να συνδυάσουμε τα σημεία 2 και 3 που θέλουμε να επισκεφτούμε ε, ή να επιλέξουμε μόνο το ένα σημείο. Είμαι ανοιχτό, λέει ο κ. Μούλντερ. Πρόεδρο, ε, οι πολιτικέ ομάδε έχουν τοποθετηθεί από αυτού. Μέχρι τώρα όχι. Ο κ. Γκάια, παρακαλώ. Κατά τη δική μου άποψη ισχύει το εξής. Όταν ε, επισκεπτόμαστε επιτόπου έργα και προγράμματα, με τον τρόπο αυτό αποκομίζουμε μία ουσιαστική εντύπωση για τις δυσκολίες που προκύπτουν. Αποκομίζουμε επίσης μια πολύ συγκεκριμένη εντύπωση πώς χρησιμοποιούνται ε, τα κονδύλια που διοχετεύονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, θα μπορέσουμε λοιπόν να αποκομίσουμε έτσι μια εικόνα ποιο είναι το πλαίσιο ασφαλείας, ε, θα μπορέσουμε να συζητήσουμε με τους άμεσα ενδιαφερόμενους κατά πόσον αντιμετωπίζουν απειλές ή κατά πόσον δέχονται εκβιασμούς για δορδοκίες Ίσως οι προσδοκίες του κυρίου Οντί να είναι υπερβολικές. Δεν νομίζω ότι θα πετύχουμε κάτι όπου να μπορούμε να πούμε ότι εδώ πράγματι πρέπει να δοθεί ε, ειδική βοήθεια για γεύματα για τα παιδιά ή για την εκπαίδευση των αστυνομικών. Μα αν συμβεί κάτι θα είναι τυχαίο και θα το λάβουμε ιδιαίτερα υπόψη μας. Αυτό που έχει σημασία είναι νομίζω θα δούμε υπό ποιε συνθήκε εργάζονται οι ανθρωπικοί και τι είδου προβλήματα απορρέουν. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω ότι είναι πιο λογικό να συνδυάσουμε δύο έργα γιατί έτσι αποκομίσουμε καλύτερη εντύπωση από το να πάμε μόνο σε ένα. Ε, έχοντας κατά νου όλα αυτά που σας είπα, εγώ είμαι υπέρ του συνδυασμού δύο ε, σημείων να επισκεφτούμε. Η κυρία Γκρέσλε. Ε, μικρόφωνο παρακαλώ. Όχι, δεν θα μιλήσει η κυρία Γκρέσλε. Ο κύριος Μούλντα. Κοιτάξτε, ε, λαμβάνοντας υπόψη αυτά που είπε ο κύριος Γκάια, προτείνω να επισκεφτούμε το δεύτερο έργο και να το συνδυάσουμε με το τρίτο. Το δεύτερο και το τρίτο εκτελούμενο έργο. Ε, πολύ ωραία λέει ο πρόεδρος. Ε, εντάξει, αυτό θα γίνει. Κλείνει και το θέμα με την IT και πάμε τώρα στο επόμενο θέμα που είναι ε, το πρώτο θέμα σε μια νέα διαδικασία. Αυτό μου το επισήμανε ο κύριος Καστήλιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, αυτές τις ε, ειδικέ εκθέσεις ε, σωστά αυτές θα εξετάζονται με μεγαλύτερη προσοχή στο μέλλον στην Ολομέλεια. Αυτή η ειδική έκθεση αφορά την αποτελεσματικότητα της αλίας. Η συγγήτρια είναι η κυρία Αντρεάσεν και εκ μέρους ε, του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου ε, θα ήθελα να καλωσορίσω τον κύριο Λάζαρο Λαζάρου και θα ήθελα ε, να του δώσω νομίζω και το λόγο. Κύριος Λαζάρου έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε και αγαπητά μέλη της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμών, ε, Είμαι στην ευτυχή θέση να σας παρουσιάσω την ειδική έκθεση παριθμών 12 του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την ε, προσαρμογή του ε, αλληλευτικού στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις πραγματικές δυνατότητες. Αυτή τη στιγμή η έκθεση υποβάλλεται σε μια κρίσιμη στιγμή της αλληλευτικής πολιτικής γιατί οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για νέα αλληλευτική πολιτική ε, πρόκειται να εξεταστούν από τις νομοθετικές αρχές. Πολύ σύντομα λοιπόν θα δω λιγάκι το υπόβαθρο της έκθεσης ε, και μετά θα επισημάνω τα βασικά συμπεράσματα και τις ε, συστάσεις του ελεγκτικού συνεδρίου. Για πάρα πολλά χρόνια ε, τα αλληλευτικά αποθέματα της Αλληλευτικής Ένωσης βρίσκονται σε φθήνουσα εξέλιξη. Η αλληλεία απειλείται απειλούνται και τα αποθέματα ε, και γενικότερα η επιβίωση του τομέα. Μετά την τελευταία προσαρμογή της ελευτικής πολιτικής το 2002 τα αλλιεύματα έχουν περιοριστεί κατά 2 εκατομμύρια τόνους ε, και περίπου 70.000 θέσεις απασχόλησης στον ελευτικό τομέα έχουν χαθεί. Όσον αφορά την αποτελεσματικότητα του αλληλευτικού στόλου, η αποτελεσματικότητα αυτή ε, θεωρείται ένας από τους σημαντικούς λόγους για την υπεραλία και για τη μείωση των αλληλευτικών αποθεμάτων. Για πάρα πολλά χρόνια με την αλληλευτική πολιτική ε, κατεβλήθησαν προσπάθειες ε, να περιοριστεί η ε, να υπάρχουν συγκεκριμένοι περιορισμοί που να επιβάλλονται στα κράτη-μέλη. Όμως, τα μέτρα τα οποία ελήφθησαν μέχρι τώρα ε, δεν απέδωσαν. Και αυτό αναφέρεται στην Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής το 2009 που περιλαμβάνει και τις ε, τρέχουσες προτάσεις. Επίσης το συνέδριο τοποθετήθηκε σε προβλήματα που έχουν σχέση με την υπερελίευση. Το έκανε αυτό σε παλαιότερες εκθέσεις και το έκανε και πιο πρόσφατα στην ειδική έκθεση υπαριθμών 7 του 2007 αλλά και σε άλλη ειδική έκθεση το 93. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε υφίστανται εδώ και πολύ καιρό. Γνωρίζοντας ότι ε, πρόκειται να τροποποιηθεί η αλληλευτική πολιτική, το ελεγκτικό συνέδριο αποφάσισε να εξετάσει τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση της υπερεαλίευσης. Εξετάσαμε τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να προσαρμοστεί η δυνατότητα των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πραγματικά αποθέματα. Τα επτά κράτη-μέλη που επισκέφθηκαμε, Δανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Πολωνία, Πορτογαλία και Ηνωμένο Βασίλειο, από κοινού αυτά ε, αντιστοιχούν, τους αναλογεί το 70% των αλληλευτικών αποθεμάτων και 80% της ε, χρηματοδότησης ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έτσι έχουμε έτσι μια σφαιρική εικόνα του τι συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Α δούμε λιγάκι ποια είναι τα βασικά μα συμπεράσματα. Το ελεγκτικό συνέδριο κατέληξε συμπεράσματα σε δύο βασικέ κατηγορίε. Το πρώτο συμπέρασμα αφορά το πλαίσιο για τη μείωση τη υπεραλίευσης και το δεύτερο αφορά το σχεδιασμό και την εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων για τη μείωση τη ε, υπεραλίευσης. Υπάρχουν τρία βασικά σημεία που θέλουν επισημάνω σχετικά με το πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται η πολιτική. Πρώτον, ε, δεν μετριέται σωστά η ε, αλίευση και υπεραλίευση. Τα μέτρα μετρούν τα σκάφη σε σχέση με το μέγεθος. Όμως εκεί δεν λαμβάνεται υπόψη η τεχνολογική πρόοδος στις αλληλευτικές μεθόδους. Ενώ η ονομαστική αξία του στόχου ε, αυξάνεται, η ικανότητα των σκαφών ε, αυξάνεται μόνο κατά 3% σε τήσια βάση. Και αυτό υπολογίστηκε από το συνέδριο γιατί διαπιστώθηκε ότι υπάρχει μια αύξηση 60% σε 16 χρόνια μέχρι το 2008. Εξάλλου, η τελευταία φορά που μετρήθηκε η ικανότητα του στόλου ήταν πριν από 15 χρόνια. Τότε υπολογίστηκε σε 40% αύξηση μετά την τελευταία έκθεση. Είναι λοιπόν πολύ δύσκολο να οριστούν οι σωστοί στόχοι για μείωση. Δεύτερον, ε, τα ανώτατα όρια της ικανότητας ε, του στόλου, ε, αυτά πλέον δεν λαμβάνονται υπόψη. Η πολιτική ορίζει τα ανώτατα όρια με βάση το μέγεθος και την ισχύ των αλληλεκτικών στόχων. Όμως τα ανώτατα όρια δεν είναι σημαντικά γιατί σας είπα το μέγεθος του στόλου είναι κάτω από τα ανώτατα όρια και μάλιστα ο στόλος ε, μπορεί να είναι κατά 200.000 μεγαλύ, τόνους μεγαλύτερους και παρόλα αυτά ανακαλύπτονται οι κανόνε. Το τρίτο που θέλω να πω είναι η αντιμετώπιση των ελληνικών δικαιωμάτων. Η ελληνική πολιτική δεν έχει σαφεί κανόνε για την αντιμετώπιση των αλληλευτικών δικαιωμάτων όταν διαλύονται τα αλληλευτικά σκάφη. Μάλιστα η αλληλευτική πολιτική είναι αντιφατική επί του θέματο. Ο βασικό κανονισμό του Συμβουλίου από το 2002 προβλέπει την απόσυρση αλληλευτικών δικαιωμάτων για τα σκάφη σκάφη που διαλύονται, όμως οι κανονισμοί ε, θέτουν ε, ετήσιες ποσοστώσεις και επιτρέπουν σε ορισμένες περιπτώσεις τα ε, δικαιώματα αυτά να μεταβιβάζονται. Ορισμένα κράτη-μέλη επιτρέπουν σε αλληλείς να πουλάνε τα δικαιώματά τους. Η πώληση των αλληλευτικών δικαιωμάτων διαλυμένων σκαφών δίνουν ένα επιπρόσθετο εισόδημα στους αλείς για να, ως ισοδύναμο μέτρο οι κανονισμοί της ελεκτικής πολιτικής δεν αναφέρουν πώς πρέπει να αντιμετωπίζονται αυτές οι περιπτώσεις ε, της πώληση των αλληλεκτικών δικαιωμάτων όταν διαλύεται ένα σκάφος. Και αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία, η ε, μεταβίβαση των δικαιωμάτων δεν διευκρινίζεται στην κοινή ελεκτική πολιτική. Ε, τα δικαστήρια αναφέρουν ότι η Νορβηγία και η Δανία έχουν προσαρμόσει την ικανότητα του στόλου χωρίς να καταφεύγουν στο εργαλείο της μεταβίβασης των ελευτικών δικαιωμάτων. Το δικαστήριο θεωρεί ότι ε, το θέμα των δικαιωμάτων πρέπει να διευκρινιστεί και να ξαχθούν τα απαραίτητα μαθήματα. Επιπλέον, θα ήθελα να αναφέρω και μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη που προετοιμάστηκε το 2010 για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τίτλο «Εργαλεία για τη διαχείριση της ελληνική πολιτικής». Και εκεί εντοπίζονται παρεμφερεί θέματα με αυτά που αναφέρουμε και εμείς στην έκθεσή μας. Υπάρχουν 7 σημεία που θέλω να επισημάνω όσον αφορά σε συγκεκριμένα μέτρα για να μειωθεί η υπεραλίευση. Πρώτον, υπάρχουν καθυστερήσεις ε, στην εφαρμογή ε, της χρηματοδότησης των κρατών μελών. Μέχρι τα τέλη του 2010, μόνο 645 εκατομμύρια, δηλαδή 15% των διαθέσιμων από τα 4,3 δις χρησιμοποιήθηκαν. Δεύτερον, τα λειτουργικά προγράμματα και οι στόχοι των κρατών μελών για τη μείωση της υπεραλίευσης δεν διευκρινίστηκαν επαρκώς. Επίσης υπήρξαν προβλήματα με προγράμματα προσαρμογής των αλληλευτικών προσπαθειών και αυτός είναι ο βασικός μηχανισμός για να αντιμετωπιστεί η χρηματοδότηση των αλληλευτικών σκαφών. Απαιτείται ε, ο καθορισμός στόχων και περιεχομένου. Αυτό όμως δεν έγινε. Τρίτον, παρότι οι επενδύσεις που ε, ενισχύουν την αλληλευτική ικανότητα είναι δημόσια η χρηματοδότηση, αυτό τελικά δεν συμβαίνει. Εμεί πιστεύουμε ότι μπορούν να γίνουν κάποιε επενδύσει έτσι ώστε τα ελεκτικά σκάφη να λεύουν ταχύτερα. Ε, τέταρτον, ε, το μητρό του Ευρωπαϊκού Ελευτικού Στόλου δεν ε, προσαρμόστηκε, δεν περιλαμβάνει τα σκάφη που διαλύθηκαν με χρηματοδότηση και ενίσχυση. Πέμπτον, ενώ από το 2003 μέχρι το 2009 είχαμε 5.800 σκάφη που ισοδυναμούν σε 350.000 ε, περίπου τόνους διαλύθηκαν με βάση το μητρό. Παρόλα αυτά η επιλογή των σκαφών ε, για διάλυση δεν ήταν στοχευμένη. Και αυτό οδήγησε στο να διαλυθούν σκάφη που δεν επηρέασαν καθόλου τα στοχευμένα αλευτικά αποθέματα. Και σε μερικές περιπτώσεις δόθηκαν ε, ενισχύσεις για σκάφη που ήταν ήδη αδρανή ή για σκάφη που εξακολουθούσαν να αλλιεύουν. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρόσφατη πρότασή της για το νέο λεπτικό ταμείο καταλήγει στο ότι να αντιμετωπίζεται η ε, υπεραλήψη μέσω της ε, διάλυσης πλέον αυτό αποδεικνύεται αναποτελεσματικό παρότι 1,7 δις ευρώ έχουν δαπανηθεί για αυτό το συγκεκριμένο μέτρο. Έκτο, ο κανονισμός ε, περί της ε, κρίσης ε, των καυσίμων είχε ανικανοποιητικά αποτελέσματα. Ο κανονισμός αυτός είχε ως στόχο να υπάρχει μεγαλύτερη διάλυση πλοίων, εξυγχρονισμός του στόλου και αυτό ως απάντηση στην κρίση του 2008. Το δικαστήριο διαπίστωσε ότι ορισμένα κράτη-μέλη ερμήνευσαν αυθαίρετα τη σχετική νομοθεσία και δεν προέβησαν σε εξοικονομίες. Παραδείγματος χάρη έμεση κρατική χρηματοδότηση για την εισαγωγή αλληλευτικών σκαφών. Δόθηκαν τέτοιου είδους ενισχύσεις. Και τέλος το δικαστήριο ε, διαπίστωσε ότι οι κανόνες ε, που ισχύουν για τα κράτη-μέλη για να αναφέρουν τα κράτη-μέλη τον περιορισμό της υπεραλήψης, αυτοί οι κανόνες είναι ανεπαρκείς και τα κράτη-μέλη ε, δεν χρησιμοποιούν τις κατευθυντήριες γραμμές Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι αδύνατο να έχει κανείς αξιόπιστες πληροφορίες ε, σε ευρωπαϊκό κοινοτικό επίπεδο. Τώρα, τι συστήνει το δικαστήριο η έκθεση συστήνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει υπόψη της ε, το κατά οι πρωτοβουλίες ε, και το όραμα ε, για τον βασικό κανονισμό είναι απαραίτητα έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερος ορισμός της υπεραλήψης και της αλληλεπτικής δραστηριότητας. Να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για να περιοριστεί η υπεραλήψη, ε, οριστούν τα όρια, να βελτιωθεί το πρόγραμμα ε, των προσπαθειών, να διευκρινιστεί το πρόγραμμα για τη μεταφορά αληφτικών δικαιωμάτων, νέες ενισχύσεις για τον εξυγχρονισμό των σκαφών, να βελτιωθεί το μητρό και να αναφέρονται οι προσπάθειες που καταβάλλονται έτσι ώστε να υπάρχει προσαρμογή της αλήψης ε, στα αποθέματα. Η έκθεση αναφέρει ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να προσφέρουν έγκαιρα χρηματοδότηση και να ε, διασφαλίζουν ε, ότι δεν θα αυξηθεί η αλληλευτική δραστηριότητα. Το Μητρό να ε, παραμένει επίκαιρο, να υπάρχει καλύτερη στόχευση και να βελτιωθούν οι προσπάθειες αναφοράς της υπεραλήψης. Τελειώνοντας θέλω να πω, το μήνυμά μας είναι η αλληλευτική πολιτική δεν θα μπορέσει να επιτύχει αν δεν περισσεί το πρόβλημα της υπεραλήψης. Και εδώ περιλαμβάνεται ο εντοπισμός του μεγέθους της υπεραλήψης, ο σχεδιασμός μέτρων για να περιστεί αυτή και η σωστή αναφορά περί της δραστηριότητας. Το δικαστήριο πιστεύει, το ελεγκτικό συνέδριο πιστεύει ότι οι προσπάθειες που καταβάλλονται προσφέρουν μια δυνατότητα ευκαιρία στις νομοθετικές αρχές για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την υπεραλήψη και είμαστε ικανοποιημένοι όπου το ελεγκτικό συνέδριο μπορεί και αυτό να συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση. Και προς ενημέρωσή σας να σας πω ότι προσκληθήκαμε από την Επιτροπή Αλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να παρουσιάσουμε αυτή την έκθεση στις 21 Μαρτίου. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και τώρα βεβαίως είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω ερωτήσεις. Ευχαριστώ κύριε Λαζάρου για την παρουσίαση της έκτακτης εκθέσεως. Όπως είπατε, η νέα διαδικασία για τις έκτακτες εκθέσεις θα ενισχύσει την ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα βοηθήσει αν και οι άλλες, Ευρωπαϊ... Ε, και οι άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές ασχολούνται με τα ίδια θέματα. Τώρα θα δώσω τον λόγο στην εισηγήτρια, την κυρία Αντρεάσεν, για να τοποθετηθεί και θα επισημάνω μόνο ότι το σχέδιο της εκθεσεώς της προβλέπεται να κατατεθεί στις 23 Τετάρτου εδώ στην Επιτροπή μας για να συζητηθεί ή τα δε συμπεράσματα της εισηγητρίας θα υπησέλθουν στο, στην έκθεση απαλλαγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κύριε Ανδρέας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Διερωτώ με ορισμένε φορές όταν ε, παρακάθιμε εδώ στην ε, ε, Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού πότε θα ξεσηκωθούν τα μέλη και θα πούν φτάνει πια με τα σφάλματα. Εδώ για την κοινή αλληλευτική πολιτική είναι από τις χειρότερες ε, εκτιμήσεις, αποτιμήσεις που έχω διαβάσει ποτέ. Εκατομμύρια, δισεκατομμύρια έχουν ε, καταβληθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την κοινή αλληλευτική πολιτική. Τι λέει τώρα η έκθεση. 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ κατασπαταλήθηκαν από το 2002 για τον παροπλισμό σκαφών χωρίς ε, να υπάρχουν πραγματικά αποτέλεσματα. Πάνω από 90% των αλλιευμάτων υπεραλλιεύονται και πέραν των βιολογικών ορίων αντοχής. Πάνω από 100.000 θέσεις απασχόλησης έχουν χαθεί στην αλλιευτική βιομηχανία η μελλοντική βιωσιμότητα της αλληλείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να εξασφαλιστεί. Η κοινή αλληλευτική πολιτική δεν ανταποκρίθηκε στις ανάγκες, δεν επέλυσε τα προβλήματα, δεν υπάρχει ενημέρωση των ε, μητρών των αλλήλων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει λάβει αποτελεσματικά μέτρα για την παρακολούθηση της κατάστασης. Η έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου επισημαίνει τα όσα ήδη γνωρίζουμε για την κοινή αλληλευτική πολιτική, ότι πρόκειται δηλαδή για απόλυτη αποτυχία. Έχει αντικαταστήσει υγιείς εθνικές πολιτικές και αντικαταστάθηκε από ένα σύστημα free for all που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν καταφέρνει να ελέγξει. Αυτή η αποτυχία λοιπόν έχει οδηγήσει και τη καταστροφή των αλλιευμάτων για παράδειγμα με ε, το να πετάγονται τα υπεραλλιεύματα στη θάλασσα είναι άλλη μία απόδειξη της αποτυχίας της ε, αλληλευτικής αυτής πολιτικής. Ποιος επέτρεψε αυτές τις πρακτικές. Η Κομισιόν μόνο υπόσχεται μεταρρύθμιση μετά από τα σχόλια του ελεγκτικού συνεδρίου. Για μένα αλλά και για πολλούς ψαράδες που έχω συνομιλήσει μαζί τους η δυσκολία είναι ότι δεν έχουμε πλέον ουδεμία εμπιστοσύνη στα πρόσωπα αυτά τα οποία δημιούργησαν την πολιτική αυτή ότι θα μπορέσουν τώρα να την αλλάξουν. Για μένα η αλλαγή είναι η, λύση είναι ξεκάθαρη. Θα πρέπει να επανεθνικοποιηθεί η ελληνική πολιτική. Εάν η έκθεση αυτή δεν μας κάνει όλους να σηκωθούμε επιτέλους και να δούμε τι γίνεται όπως το βλέπουν οι ε, συντάκτες εκθέσεως, δεν θα μείνει δηλαδή αλληλευτική ε, βιομηχανία για πολύ καιρό. Θα θέσω ορισμένε ερωτήσει τώρα στο Ελεκτικό Συνέδριο αλλά και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το Συνέδριο γνωρίζει συγκεκριμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένε χώρε μέλη, ότι δηλαδή δεν έχουν κάνει του ελέγχου όπω Κύπρο, Ελλάδα και Ολλανδία. Η Κομισιόν το 2011 κατέθεσε σχέδια για την τροποποίηση της αλληλευτικής πολιτικής μετά από τα σχόλια του ελεγκτικού συνεδρίου πότε θα πρέπει να καταθέσει τα σχέδια μεταρρυθμίσεων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όταν λέει το ελεγκτικό συνέδριο ότι οι χώρες μέλη θα πρέπει, θα πρέπει, σημαίνει αυτό ότι θα επιβληθούν αυτομάτως κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Για τη δεύτερη τώρα σύσταση προς τις χώρες μέλη. Δεν είναι αντίθετο με τα ένστικτά τους ε, να λένε ότι η βελτίωση των σκαφών δεν θα αυξήσει την αλληλευτική τους ικανότητα και γιατί δεν τίθενται επιτέλους τα αναγνωρισμένα προβλήματα επιτάπητος. Τώρα, η Κομισιόν, γιατί η τελευταία σας αξιολόγηση της υπερικανότητα, τη προορικής ικανότητα αλίευσης των σκαφών έγινε πριν από 15 χρόνια. Οι περισσότερες χώρες μέλη δεν συντάσσουν επαρκεί εκθέσεις. Αλλά είμαι βέβαιο ότι στο κτίριο Μπορσέτ οι σχετικέ ε, ομάδε επιρρογνωμόνων συναντώνται αρκετά συχνά. λοιπόν η εκπρόσωποι των Υπουργείων κάνουν τίποτα άλλο εκτός από το να συνομιλούν απλά όταν έρχονται εδώ στις Βρυξέλλες. Αυτά ήταν λοιπόν για την ώρα τα ερωτήματά μου. Ευχαριστώ κύριε Συγήτρια και πριν δώσω τον λόγο στους εκπροσώπους της Κομισιόν θα ρωτήσω πρώτα τα μέλη της Επιτροπής εάν έχουν άλλες ερωτήσεις είτε προς το Ελεγκτικό Συνέδριο είτε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εσείς κύριε Γκάιερ. Πρώτη ερώτηση είναι διαδικαστική. Είπατε, εισάγοντας το θέμα, ότι η έκθεση Αντρεάσεν θα, αποτελε... θα συναποτελέσει ειδικό για την απαλλαγή. Οι σύμβουλοι της πολιτικής ομάδας μου είπαν ότι είναι η πρώτη έκθεση η οποία θα μπει σε μια νέα διαδικασία εφόσον δηλαδή θα γίνει μια πλήρης έκθεση η οποία θα ψηφιστεί και από μόνη της θα αποτελέσει τη γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εγώ νομίζω ότι εδώ υπάρχει κάποια διαφορά ανάμεσα σε αυτό που έχω κατανοήσει και σε αυτό που εξήγησατε εσεί και γι' αυτό θέλω να ρωτήσω και πάλι για να είμαστε βέβαιοι σχετικά με την διαδικασία. Ίσως είναι δυνατόν λοιπόν εν προκειμένου να λάβουμε κάποια περισσότερη ενημέρωση για τους συναδέλφους διότι πρόκειται και μια τροποποίηση του τρόπου εργασίας της Επιτροπής μας που μέχρι τώρα δεν έχουν ψηφιστεί ε, οι γνωμοδοτήσεις μας για τις εκθέσεις του ελεγκτικού συνεδρίου. Έχουμε ορίσει συγητή και έχουμε συζητήσει. Και ο εισηγητής της απαλλαγής της Κομισιόν είχε το ελεύθερο να την περιλάβει η γνωμοδότηση αυτή ή όχι. Λοιπόν, θέλω τώρα εδώ να διευκρινιστεί πρώτα αυτό, να υπάρχει ασφάλεια δηλαδή επί του θέματο και να δούμε πώ θα προχωρήσει η διαδικασία. Αν δηλαδή θα ψηφίσουμε τελικά την έκθεση Αντρέα ή όχι. Επειδή της ουσίας, όντως είναι πραγματικά τρομακτικά τα όσα μας ανακοινώνει το ελεγκτικό συνέδριο και τα εξήγησε αυτά και η κυρία Αντρεάσεν, θέτοντας την ερώτηση πότε πια θα πούμε φτάνει πια για λογαριασμό των σοσιαλδημοκρατών μπορώ να πω ότι χαιρόμαστε που η Κομισιόν αρχίζει να αποστασιοποιείται από την, από εφαρμογή του προγράμματος αυτού διότι αυτά που λέει το ελεγκτικό συνέδριο για την εκτέλεση του προγράμματος είναι τέτοια που πραγματικά ε, οδηγούν στην ανάγκη εκβάθρων αναθεώρησης. Οι δε συντονιστέ της πολιτικής μου ομάδας στην Επιτροπή Αλίας μου λένε ότι θα ζητήσουν από την Επιτροπή να μην προχωρήσει στην εφαρμογή του προγράμματος. Και αυτό ενδεχομένως να εγκριθεί και από την πλειοψηφία της ε, Επιτροπής Αλίας. Ίσως λοιπόν όντως να οδηγηθούμε εδώ σε ένα πέρας. Πρόεδρος. Ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχουν ε, άλλε παρατηρήσει. από ό,τι φαίνεται αυτή τη στιγμή. Δεν επιθυμεί κανεί άλλο το λόγο. Κοιτάξτε, οι δικές μου οι παρατηρήσεις για τη διαδικασία αφορούν ε, την τοποθέτηση στο Continuous. Ε, και πράγματι ισχύει αυτό που είπατε κύριε Γκάια, αγαπητέ συνάδελφε, ότι εδώ συζητάμε για ε, σχέδιο έκθεση της κυρίας Αντράσεν. Θα συμφωνήσουμε για τις ε, τροπολογίες και μετά θα κάνουμε με την έκθεση αυτή ό,τι κάνουμε και με τις υπόλοιπες εκθέσεις. Βεβαίως πρέπει να πω ότι τα συμπεράσματα που θα προκύψουν για αυτήν την έκθεση θα παίξουν ρόλο στην διαδικασία απαλλαγής. Θα υπάρξουν δηλαδή ε, επιπτώσεις και προς τις δύο κατευθύνσεις. Ε, πολύ ωραία. Και θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο ε, στην εκπρόσωπο της Κομισιόν ή στου εκπροσώπους είναι ο κύριος Πένασλάντο και ο κύριος Τζόνσον. Δεν ξέρω ποιος επιθυμεί να τοποθετηθεί. Παρακαλώ. Thank you, Chairman. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς να σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί πάρα πολύ θετική την έκθεση του Ελληνικού Συνεδρίου και όσον αφορά τον χρονισμό και όσον αφορά το περιεχόμενο όπως ελέγχθη είναι ακριβώς ό,τι πρέπει για την ε, προβληματική που έχει αναπτυχθεί όσον αφορά την μεταρρύθμιση της κοινή ελευθερικής πολιτικής. Θεωρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι αυτό το πρόβλημα της ε, υπερπαραγωγής στην Ευρώπη ή της τελικά το τι θα κάνουμε θεωρείται... Ε, ε, μόνο έτσι, έτσι, θα βγάλουμε άκρη με τη μεταρρύθμιση και θα πρέπει να λάβει υπόψη τις συστάσεις του ελεκτικού συνεδρίου. Για να δούμε τώρα, να σα πω τι πρεσβεύουμε εμεί όσον αφορά τα επιμέρους στοιχεία που αναφέρθηκαν. Ναι, συμφωνούμε όσον αφορά την υπεραλίευση. Έχουμε στατικές παραμέτρους που όμως δεν καλύπτουν αυτά που θέλουμε όσον αφορά τη σύλληψη του προβλήματος. Γιατί δεν είναι στατικό πράγμα η υπεραλίευση. Η υπεραλίευση υπάρχει διότι έχουμε συνεχή τεχνική και τεχνολογική πρόοδο όσον αφορά την αλίευση, οπότε όλο ένα και περισσότερο μπορούν οι ελευτικοί στόλοι να αλίευουν περισσότερα πλοία. Επομένως πρόκειται για κάτι που οι στατικές παράμετροι δεν μπορούν ποτέ να υπολογίσουν. Επίσης συμφωνούμε με το ότι όσοι έχουν σήμερα τα, τα, οι οροφές δεν αρκούν. Έχουμε σήμερα ονομαστική τήρηση των ε, ορφών όπως ε, αναφέρονται από τις στατικές παραμέτρους αλλά ούτε αυτό είναι ικανό να καλύψει το πρόβλημα όσον αφορά την ανάπτυξη, την, τις δυνατότητες της των στόλων για αλίευση. Τώρα, Όντω χρειάζεται περισσότερη σαφάνεια, είναι πάρα πολύ σημαντικό τώρα να δούμε τι γίνεται όσον αφορά τα δικαιώματα μεταβίβασης ε, για να δούμε τι γίνεται με τα επίπεδα λήψη. Πάντως, ό,τι και να γίνει με τα δικαιώματα, συμφωνούμε ότι η κατάσταση άλλος έχει όσον αφορά το κάθε κράτος μέλος. Και ό,τι και να γίνεται όσον αφορά τα δικαιώματα, αυτό με τίποτε δεν αυξάνει το πόσο δικαιούται να κάθε κράτος μέλος, το οποίο κάθε φορά αυτό εξαρτάται από την πολιτική διατήρηση και προστασία των λευτικών πόρων. Αυτό καθορίζει τι δικαιούται κάθε κράτος. Αφήστε που υπάρχει και κάποιο είδου σύγχυση, κάποια κρατημέλη σε το πώ γίνεται η μεταβίβαση των ε, ε, δικαιωμάτων. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σχέση με την αύξηση των ε, δυνατοτήτων αλίευσης. Και νομίζω ότι πάρα πολύ ε, πρέπει να ληφθεί υπόψη το ότι το Ταμείο έχει ολόκληρο σύστημα Και πήρε πολύ χρόνο τόσο ώστε να συγκροτηθεί αυτό το σύστημα. Και αυτά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για ό,τι ισχύσει στο μέλλον για τα ταμεία. Απλούστευση, ένταξη σε όλες τις πολιτικές και έτσι να μπορέσουμε να επιλύσουμε το πρόβλημα στο μέλλον. Επίσης, έχουμε το θέμα των ε, προγραμμάτων που παρακολουθούμε εμείς με προσοχή στις περιπτώσεις που υπάρχουν αξιώσεις ε, καταβολής που δεν πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις εμείς δεν εκταμιεύουμε μέχρι ότου ξεκαθαριστεί το πρόβλημα. Επομένως δεν υπάρχει κανένας είδους υποχρέωση ε, καταβολής στα κρατημέλη εάν δεν εκτελούνται όπως πρέπει τα προγράμματα. Άλλο. Για τις ε, επενδύσεις. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Σε σχέση με το EFF που δεν είπαμε αντιστοιχεί λόγω των, λόγω των στατικών παραμέτρων στα πραγματικά κιλοβάτ κλπ. Απευθυνθήκαμε στα κράτη-μέλη πέρυσι και είπαμε να μα πούν ακριβώ τι επενδύσεις έκαναν. Και εμείς θα κρίνουμε, είπαμε, εάν αυτές οι επενδύσεις αντιστοιχούν στην νομική υποχρέωση του να μην αυξάνεται η αελίευση. Και έτσι θα λάβουμε τις σχετικές αποφάσεις για το τι δικαιούται το κάθε κράτο μέλος. Τώρα, όσον αφορά κάποιο είδου νεολόγια και την ενημέρωσή του. προσπαθήσαμε πάρα πολύ σε κάποια μέλη να το ρυθμίσουμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πλέον ενημερώνει το μέλη και ενημερώνει τα νεολόγια. Όπου <coughs> υπάρχουν ελλείψεις, απευθύνουμε στα κρατημέλη για να ενημερώσουμε το ενοιολόγιο. Επίσης, όσον αφορά την απόσταση των πλοίων, εδώ δεν έχουμε σωστή σχέση κόστους αποτελέσματος. Και όσον αφορά την επιλογή από πλευρά κρατών μελών το ποια πλοία θα προπιστούν, δεν έχει γίνει καλή δουλειά. Και είπαμε. Θα πρέπει να γίνει περαιτέρω επεξεργασία, να είναι πιο λεπτομερείς οι προβλέψεις για το ποια πλοία θα προβληστούν κάθε φορά. Και όπως ξέρετε, σκοπεύουμε να καταργήσουμε την ε, χρηματοδότηση, επιδότηση της, ε, ε, του προβλησμού των πλοίων. Έχουμε ήδη εκδώσει καθημερινές γραμμές όσον αφορά το τι έχουν κάνει τα κράτη-μέλη για την υπεραλίευση. Προσπαθούμε να είμαστε όσο γίνεται πιο αντικειμενική, άλλα κρατημέλη τα ετήρησαν, αλλά όχι. Πάντως τελικά κάθε φορά που συμβουλευόμαστε το STCF καταλήγουμε στο να διαπιστώσουμε ότι η κατάσταση είναι πολύ περίπλοκη. Γιατί δεν αρκεί η προσαρμογή των παραμέτρων στους πόρους. Ε, πάντοτε τα κράτη-μέλη αρνούνται το πρόβλημα. Δεν μπορούμε να βρούμε ορισμό που να καλύπτει τα προβλήματα. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει το να πάυσει αυτή η παραδοσιακή πολιτική των ονομαστικών στατικών παραμέτρων που δεν μπορούν να καλύψουν τεχνικά προβλήματα και να αντικατασταθεί το σχεδόν σύστημα με ένα άλλο σύστημα να λαμβάνει υπόψη τον κλάδο και χωρίς καθυντήρηση από τις Βρυξέλλες, έτσι να καθορίζεται χωρίς ευρώ από, από την τσέπη του καταναλωτή να μας λένε τι, τι, τι θεωρούν υπεραλίευση επί τη βάση ε, της αϊφόρου αλίας. Έχουμε τώρα κάποιες ε, συγκεκριμένες ερωτήσεις να σας απαντήσω. Έχω τα εξή δύο να σας πω. Όσον αφορά την απόρριψη του ελίγματος, εμείς προτείνουμε για την απόρριψη να γίνει προσαρμογή βαθμία. Είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 3 της Συνθήκης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, κοινή αληθική πολιτική. Αυτόματες ε, κυρώσεις. Το δίκαιο κυρώσεις εμείς πάντοτε είμαστε σε ετοιμότητα σε σχέση με την επιβολή αυτών των κυρώσεων, αλλά πάντοτε θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει. Γιατί σήμερα σε σχέση με τα ταμεία δεν υπάρχει νομική βάση ή δεν μπορούμε να αρνηθούμε την επιστροφή των πόρων στα κράτη-μέλη. Ε, όμως αυτό αφορά κάποια κριτήρια επιλεξιμότητας. Θα πρέπει κάποιος να, να, να, να μην καταστεί επιλέξιμος για να μιλάει τα χρήματα. Επίσης, θέλουμε ένα καλύτερο σύστημα για να εξασφαλίσουμε την αιρεσιμότητα σε σχέση με τις δημόσιες δαπάνες. Διότι, Πρόεδρε, η πρόταση της Επιτροπής για τη μέλουσα και πολιτική αλίας θα καθορίσει και την ρεσιμότητα για τις δημόσιες σχετικές δαπάνες. Γι' αυτό και είπαμε, θα πρέπει να μας βοηθήσετε, εάν δεν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις, να μην καταβάλουμε. Βοηθήστε απλώς νομοθετικές. Τώρα, για το μέσο πρόθεσμο, ναι. Ναι. θα προχωρήσει η λειτουργία του Ταμείου Ελίας. Θα έχουμε το κείμενο το σχετικό φέτος. Πριν από 15 χρόνια ξέρετε ότι γίνεται τελευταίος υπολογισμός της υπεραλίευσης. Και αυτό γιατί, διότι τότε έπρεπε να έχουμε προετοιμάσει την τεχνική βάση που για μας αποτελεί το τι πολιτική θα ακολουθήσουμε για τα επόμενα 7 χρόνια. Το θέμα είναι κατά πόσο θα ήταν υποχρεωτική η ρύθμιση σε σχέση με την μείωση της υπερελίευση. Αυτή η πολιτική επομένω της υποχρεωτικότητας για να συσταλεί αυτή, να συγκρατηθεί αυτή η υπεραλίευση το 2002 έπαυσε από το Συμβούλιο. Και από τότε λοιπόν δεν έχουμε υποχρέωση μείωση της υπεραλίευση. Αυτά αποφάσισε το Συμβούλιο το 2002. Οπότε έχουμε τώρα το την καινούργια πολιτική. Ευχαριστώ. Yeah, thank you very much. Uh, I... Σας ευχαριστώ. Βεβαίως θα μπορούσαν να συζητηθούν ακόμη περισσότερο τα πράγματα, αλλά στις 12.30 οφείλουμε να εγκαταλείψουμε την αίθουσα. Δεν έχουμε πλέον τόσο πολύ χρόνο. Δεν ξέρω και τι να κάνουμε με την ε, συνεδρίαση των συντονιστών. Ωστόσο θα προτείνω να δώσουμε χρόνο ενός λεπτού στο ελεγκτικό συνέδριο για να απαντήσει και αν θέλει να προσθέσει λεπτομέρειες γραπτός και θα το ξανασυζητήσουμε και θα ψηφίσουμε ξανά στην παρούσα Επιτροπή. Ευχαριστώ κύριε, κύριε Λαζάρου λοιπόν. Για το πρώτο ερώτημα του εισηγητού σχετικά με το εάν το δικαστήριο, αν το ελεγκτικό συνέδριο γνωρίζει περί προβλημάτων στις κάτω χώρες Ελλάδα και Κύπρο, η απάντηση είναι ότι ο στόχο τη έκτακτη έκθεση ήταν να δοθεί μια συνολική επισκόπηση των προβλημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και για το λόγο αυτό επιλέξαμε ορισμένε χώρε μέλη, οι οποίε συνολικά ε, ε, αντιπροσωπεύουν το 80% του ε, προπολογισμού. Δεν έχουμε επισκεφθεί τι χώρε αυτέ, ούτε καμία άλλη άλλωστε, και δεν μπορούμε να σχολιάσουμε επί συγκεκριμένων προβλημάτων. Σε ό,τι αφορά το εάν θα πρέπει να επιβάλλονται αυτομάτω κυρώσει, Αυτό ξεφεύγει από τις αρμοδιότητες του ελεγκτικού ε, συνεδρίου. Είναι θέμα πολιτικό. Αναφέρομαι ταχύτατα στην ειδική έκθεση, στην παράγραφο 34, που λέμε ε, ότι η υποκοινή διαχείριση οι χώρες μέλη που είναι αρμόδιες για την διαχείριση, εκεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει περιορισμένη δυνατότητα να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται. Και στην παράγραφο 71 λέμε ότι οι ρυθμίσεις της κοινή αλληλευτικής πολιτικής για χώρες μέλη οι οποίες δεν έχουν συντάξει επαρκείς εκθέσεις για τους αλληλευτικούς του στόλους δεν υπέστησαν ε, κυρώσεις. Ευχαριστώ για τις σύντομες απαντήσεις σας. Εισηγείτε για ένα λεπτό. Τι να προσθέσω, δεν έχω τίποτε να προσθέσω για την ώρα. Θα συζητήσουμε αργότερα. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ όλες και όλους. Και εδώ φτάσαμε στο πέρα της σημερινή ημερησίας διατάξεως και οι επόμενες συνεδριάσεις θα διεξαχθούν σύμφωνα με τις ημερομηνίε που έχουμε ανακοινώσει 28-29 Φεβρουαρίου. Ευχαριστώ άλλωστε τους εκπροσώπους των άλλων θεσμικών οργάνων που είναι παρόντα. Θα κλείσω εδώ τη συνεδρίαση και να προχωρήσουμε ευθύ αμέσω στη συνεδρίαση των συντονιστών. Θα παρακαλέσω λοιπόν να μπορέσουμε να συνεχίσουμε το ταχύτερο δυνατό και κλεισμένο των θυρών.